την περίπτωση της Σφασιλάδης, την περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τουλάνι Μασέκο και Μπέκι Μακούμπου. Και παρακαλώ τους συντάκτες του ψηφίσματος να λάβουν το λόγο πρώτοι. Ο κύριος Μάρκ Τεμέσμεκερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. από την κατάργηση του συντάγματο και την κατάργηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων το 1973 η κατάσταση της απόλυτης μοναρχίας της Βοζιλάνδη μπορεί αντίθεση με χώρες γειτονικές όπως η Νότια Αφρική ή η Μοζαμβίκη. Και έχουμε τώρα τον βασιλέα Μσουάτη τον τρίτο, ο οποίος αρνείται να μοιραστεί την εξουσία ή να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε μια κατάσταση λοιπόν με τεράστια ποσοστά φτώχεια σημαντικά και πολύ ψηλότερα οποιοδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου ποσοστά του AIDS και μεταξύ άλλων έχουμε την καταδίκη των Τουλάνι Μασέκο και του Μπέκι Μακούμπου που δεν είναι όμως μεμονωμένες ε, περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων, το δικαίωμα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε, του, ε, κλεισίματα ή θέση εκτό νόμου συνδικαλιστικών σωματείων. Παρ' όλα αυτά όμω ο Βαζιλάνδη παραμένει μέλο τη Συμφωνία του Κοτονού και άλλων διεθνών ε, συμβάσεων οι οποίε ε, απαιτούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να αρκούμαστε μόνο στην έκκληση για απευθεία και για άμεση απελευθέρωση των δύο κρατουμένων, αλλά, για επανα... αλλά πρέπει να ζητούμε την επαναφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Χωράω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Δεμεσμάκερ, οι Μασέκο και Μακούμπου συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν μόνο και μόνο επειδή καταφέρθηκαν κατά του δικαστικού συστήματος Βαζιλάνδες. Ο ένας δικηγόρος, ο άλλος αρχισυντάκτης της μεγαλύτερης εφημερίδας της χώρας. η Σουαζιλάνδοι από την ανεξαρτησία της από το 1968 αντιμετωπίζει διαρκώς καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Έχει καθεστώς απόλυτης μοναρχίας. Παραμένει όμως μια χώρα που εντάσσεται στο σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούνται τα θερμαδικαιώματα δικαιώματα ως προκαταρκτική όρη. Αυτό ζητούμε με το ψηφισμό μας. Κατά τα μας φαίνεται Προφανέ ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρούμε σχέσει με εκείνου που συστηματικά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε ότι το ψήφισμά μα θα απευθύνει ένα σαφέ και απερίφραστο μήνυμα στην ε, κυβέρνηση τη Βασιλάνδη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χόιμπους. Χόιμπουχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο Τουλάνι Μασέκο και ο Μπέκι Μακούμπου ήθελαν να, καταστήσουν, ήθελαν να προσελκύσουν την προσοχή ως προς τη χώρα τους για τα δικαιώματα και το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις που έχουν επαναληφθεί πολλές φορές. Υπάρχει μια προσπάθεια ε, εκφοβισμού των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κρατικές δομές και τα όργανα της Βαζιλάνδης ε, πρέπει να σεβαστούν το ίδιο τους το Σύνταγμα του 2005, εκεί όπου υπάρχει δυνάμει του άρθρο 24 η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των ασωμαζικής ενημέρωσης. Ε, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να σεβαστούν και τις διατάξεις της Συμφωνίας του Κοτονού με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε και οι δύο κρατούμενοι να αποφυλακιστούν αμέσως, αλλά όχι μόνο αυτοί. Οποιοδήποτε άλλος έχει φυλακιστεί στο Ασυλάνδη για αντίστοιχους λόγους. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τους όρους φυλάκισης, γιατί βρίσκονται σε απομόνωση και αυτό ισοδυναμεί με βασανισμό. Πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθύνουμε ένα σαφές και περίφραστο μήνυμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο Χαβιέρ Νάρτ τώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε. Έχουμε συνηθίσει ε, σε πολλαπλές καταδίκες, ρητορικές όμως, όπου προσπαθούμε να ε, χαϊδεύσουμε τη συνείδησή μας. Αλλά πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Έχουμε το άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης. Είναι η δημοκρατική ρήτρα που ποτέ όμως ε, δεν εφαρμόζεται παρά το ότι τα πάντα έχουν παραβιαστεί. Έχουμε τη συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 9 σημείο 2 που και αυτό έχει μια συγκεκριμένη δημοκρατική διάσταση και τη συμφωνία ε, σύνδεσης με χώρες μεταξύ των οποίων είναι και η Σουαζιλάνδια από τις οποίες απαιτείται δημοκρατική συμπεριφορά και πρέπει να απαιτήσουμε πραγματικά ε, στην πράξη τη δημοκρατική συμπεριφορά. Βαρέθηκα τι καταδίκε και πρέπει να είναι απερίφραστο το μήνυμά μα ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία ή προτίμηση κανενό είδου εάν δεν σεβαστούν οι χώρε τι συμφωνίε, ε, τι δημοκρατικέ ρήτρε και τι δημοκρατικέ απαιτήσει που περιλαμβάνουν οι συμφωνίε μα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Η Λίδια Σέντρα Ροντρίγκεθ τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Σουαζιλάνδη είναι μια περίπτωση παραβίασης της ε, ελευθερίας έκβασης συνεταιρίζεστε, συνέρχεστε, παραβιάζονται και τα δικαιώματα συμμετοχής ε, των εργαζομένων σε συνδικάτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ίσως αυτό για τις πολυεθνικές. Όλα αυτά τα δικαιώματα ε, είναι κατοχυρωμένα στην ε, Οικουμενική Διοίκηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το Κοινοβούλιο λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είμαστε άτεγκτοι και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μηχανισμό έχουν στη διάθεσή μας ώστε η κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης να εγγυηθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων ε, και των αγροτών καθώς και την ελευθερία έκφρασης, τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό πληθυσμό. Επίσης, Θέλουμε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ποιότητα, στο ποιόν αν θέλετε τη δημοκρατία σε κάποια κράτη-μέλη όπως στην Ισπανία που έχουμε έναν νόμο φήμωσης ε, των ε, μέσων ενημέρωσης, στη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, βασανιστήρα, κρατήσεις, ε, βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας, φυλάκιση συνδικαλιστών, ε, πρέπει ε, να αγωνιστούμε για την ελευθερία και στα δικά μας κράτη-μέλη, γιατί τέλος θα, μας, ε, θα είμαστε αξιόπιστοι σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλαμ για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση των Ευρωπαίων Δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη ήταν προβληματική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ε, το πούμε μετριοπαθή τρόπο. Έχει όμως επιδεινωθεί δραματικά ε, και σήμερα έχουμε ε, την περίπτωση ε, του δικηγόρου του Λάνη Μασέκο, ο οποίος προσπαθήσει να υποστηρίξει ε, τα δικαιώματα συνδικαλιστική οργάνωση και έχουμε και ε, τον αρχισυντάκτη τη μόνη ανεξάρτητη εφημερίδα τη χώρα ε, Μπέκη Μακούμπου, οι οποίοι αμφότεροι με γελίε ποινέ για περιφρόνηση δικαστηρίου καταδικάστηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη πρέπει να γίνεται σεβαστή ανα πάσα στιγμή. Και ζητούμε από τις αρχές της ε, Σουαζιλάνδης ε, να απελευθερώσουν ε, ανεφόρον αυτά τα δύο άτομα αλλά και οποιονδήποτε άλλο ο οποίος καταδικάστηκε επειδή έκανε χρήση του της ελευθερίας έκφρασης. Ζητούμε από τη Σουαζιλάνδη ανεφόρον να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως υποκύπτει και από τη Συμφωνία του Κοτονού που περιλαμβάνει την ελευθερία έκφρασης. Το να δίνουμε προτιμήσεις στη Σουαζιλάνδη ε, πρέπει να σχετιστεί με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από την τοπική κυβέρνηση. Η Συνομοσπονδία Συνεργαστικών Οργανώσεων ε, δεν είναι πλέον παράνομη από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα πρώτο βήμα όμως αυτό. Ελπίζουμε στη ίδια κατεύθυνση να συνεχίσει η χώρα. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mrs. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μαζικές οι πολιτικές καταστολές, κλίμα φόβου ε, στη χώρα. Η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται τη στήριξή μας κατεπηγόντως. Ε, και σίγουρα τα συνδικαλιστικό κίνημα είναι σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ε, πρέπει να δώσει ε, την απαραίτητη σημασία. Και λέμε με αυτό το ψήφισμά μα ε, στην κυβέρνηση τη Σουαζιλάνδη ότι εμεί προσέχουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ρασιακών δικαιωμάτων και η κράτηση του Μασέκο και του Μακούμπου είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα ανεφόρων. Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε όσου μάχονται για την πρόοδο στη Ζουαζιλάνδη και αυτό θα πρέπει να το ε, ε, συντεριάξουμε και με πράξη και όχι να μένουμε στα λόγια. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να βοηθήσουμε στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πράξει τα δέοντα και εκπρόσωποι τη στη Σουαζιλάνδη. Κύριε Επίτροπε, οι ΙΠΑ έχουν δράσει. Εμεί γιατί όχι. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπο πολιτικών ομάδων τώρα έχουν το λόγο με πρώτον εκ μέρους του ΕΛΚ, τον Κέλλη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η περίπτωση της Σουαζιλάνδης ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Οποιαδήποτε χώρα η οποία δηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1973 και ισχύει 42 χρόνια μετά, αυτό μιλάει από μόνο του. Και αυτό ισχύει και για τα, τους δύο ανθρώπους αυτούς, τους κυρίους Μασέκο και Μακούτμπου, και ο δικαστής επικεφαλής του δικαστηρίου ε, είχε υποστεί επικρίσεις από την εφημερίδα του ε, Μακούμπου και αυτό δείχνει πόσο ε, υπάρχει και κατά πόσο υπάρχει ελευθεροτυπία. Στο δεύτερο ήμιση του έτους θα έχουμε μια επίσημη επίσκεψη από εκπροσώπους της χώρας και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχει αρθεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και έχουν απελευθερωθεί οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να προσυπογράψουμε καμία συμφωνία. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γιονγκέριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το πέρσι τον Αυγουστό, ο Πρωθυπουργός της Σουαζιλάνδης ε, μίλησε για την ε, αφαίρεση λόγου από δύο ε, υπέρμαστον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το, τη διάσκεψη κορυφής της Ουάσιγκτον και παρά αυτά τα γεγονότα δυστυχώς συμμετέχει στο ε, πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας και έχει προτιμησιακό καθεστώς μέσα στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αποτροπιαστικές πράξεις και παραβιάσεις της ε, κυβέρνησης της Σουαζιλάντης θα πρέπει να ζητήσουμε και από τα Ηνωμένα Έθνη την ερεύνηση κατάστασης όσο αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Και θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς ε, των, ε, της προτιμησιακής βοήθειας. Τώρα είναι η, ήρθε η ώρα να δείξουμε το μαστίγιο. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, στη Σουαζιλάνδη το θέμα της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας του συνέρχεσθε έχει μεγάλη σημασία. Οι δύο αυτοί άνθρωποι προσπάθησαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και την ελευθερία του εκφράζεστε. Το 2014 καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια φυλάκισης γιατί καταδίκαζαν το καθεστώς της χώρας τους. Όπως είπε και ο συνάδελφος Κέλλη, ο δικαστής επικεφαλής της υπόθεσης είχε επικριθεί από την εφημερίδα του κυρίου Μασέκο. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να υπάρχει, έχει μεγάλη σημασία η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μαζέκο έστειλε μία επιστολή από τη φυλακή λέγοντας ότι θα πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι αυτό είναι η, η κορονίδα της αξιοπρέπειας. Ο κύριος Ντεχόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με την ε, διαπραγμάτευση και τη συμφωνία του Κοτονού, η Σουαζιλάνδη θα πρέπει να διασφαλίσει την ελευθερία του εκφράζεστε. Γι' αυτό πιστεύω ότι η φυλάκιση των Μασέκο και Μακούμπου αποτελεί κατάφορη παροβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει δικαίωμα κανένα καθεστώς να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα βίας και καταστολής. Θα πρέπει να δείξουμε στη Σουαζιλάνδη ότι δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης θα πρέπει να προωθήσει τις δημοκρατικές αξίες όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει τίποτα άλλο παρά ε, να διαφυλάσσονται αυτά τα δικαιώματα και εμείς είμαστε εκείνοι που θα εποπτεύσουμε την κατάσταση στη Σουαζιλάνδη. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να είναι εμπορικός εταίρος πια αυτή η χώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχουμε τη δικασία Καρστιάη. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, η διεθνή αλληλεγγύη να εκφραστεί προς τους πολιτικούς αντιφρονούντες που φυλακίστηκαν από το κατασταλτικό καθεστώς της Βασιλάνδης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια ενώπιον ενό τέτοιου ζητήματο που αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Αζιλάνδη έχει αυτοδεσμευτεί δύναμη τη Συμφωνία του Κοτονού να σέβεται ο κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, δημοκρατία. Ελευθερία δηλαδή έκφραση, ελευθερία μέσω μαζική ενημέρωση πρέπει να αναλάβει πλέον σαφή μέτρα η κυβέρνηση για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, ε, τη δημοκρατία, τον πλουραλισμό και ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει πλήρη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων με βάση και σύμφωνα με τις διεθνείς και εγχώριες υποχρεώσεις σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να θέτει σε κίνδυνο η Σουαζιλάνδη και το καθεστώ της, ε, καθεστώς την σωματική ακυρεότητα των ε, αντιφρονούντων. Θα πρέπει να τους απελευθερώσει το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νότης Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Σουαζιλάνδη είναι γνωστή. Εδώ και 41 χρόνια υπάρχει μια απόλυτη μοναρχία, έχει επιβληθεί κατάσταση ανάγκης δεν λειτουργεί ουσιαστικά η δημοκρατία το κράτος δικαίου και ούτε το δικαστικό σύστημα παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν συλλογικές ελευθερίες στους ίδιους τους εργαζόμενους. έχουμε λοιπόν τη συνέχεια μιας κατάστασης καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ο μασένκο εν προκειμένου είναι ένας γνωστός δικηγόρος ο οποίος υπερασπίζεται τους εργαζόμενους είναι δικηγόρος των συνδικάτων και τόλμησε να ασκήσει κριτική στο σύστημα δικαιοσύνης της χώρας του. Ο Μαγκούγκου είναι άνθρωπος που είναι δημοσιογράφος, είναι και αυτός έχει ασκήσει κριτική στο δικαστικό σύστημα. Έχουν επιβληθεί λοιπόν εξοδοτικές ποινές, πηγές, ποινές αντίθετες με την αρχή τη αναλογικότητα, Είναι δεδομένο ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ζουαζιλάνδη σύμφωνα με την συμφωνία του κοτονού πρέπει να σέβεται τη δημοκρατία όμως δεν το κάνει. επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα ενάντια σε αυτό το αντιδημοκρατικό καθεστώς. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Μασίμο Καστάλτο. κύριος Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Σουαζιλάνδη επικρατεί μία μοναρχία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μασέκο και Μακούμπο δυστυχώς διώχθησαν. Ο ένας ε, επέκρινε το δικαστικό σύστημα και ο άλλος ήταν ο τελευταίος εκδότης ο οποίος είχε μία ανεξάρτητη εφημερίδα στη Σουαζιλάνδη υπό το, γεγονό, υπό το φως του γεγονότος ότι το 40% του ΑΕΠ της χώρας το κατέχει η Coca-Cola με την παρουσία της στη χώρα μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ακόμα και η ΙΠΑ δεν αποφάσισαν να άρουν την προτιμησιακή συμφωνία το Νοέμβριο του 2014 εφόσον δεν πέρασαν οι μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της μελλοντική συμφωνίας οικονομικών εταιρικών σχέσεων δεν αποτελεί ε, κενό γράμμα. Όπως δεν είναι κενό γράμμα και το κοτονού. Θα πρέπει λοιπόν να χτυπήσουμε τη γροφιά μας στο τραπέζι όταν μιλάμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαφορετικά χάνουμε εμείς την αξιοπιστία μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ. Στην η Ιταλία υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται «Σκέρτσια πάρτε», δηλαδή δεν αστειευόμαστε. Μιλήσαμε λοιπόν για τους Βιρμανούς, για τους μετανάστες της Βιρμανίας, μα εμείς ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση από τη Λιβύη και τη Συρία και τώρα μας απασχολεί η Σουαζιλάνδη δεν ξέρω καν ξέρετε, ξέρουμε οι περισσότεροι που βρίσκεται η Σουαζιλάνδη. Πού βρίσκεται η Σουαζιλάνδη, ε, κύριοι. Ας ασχοληθούμε με τους νέους, τους ηλικιωμένες, με το μέλλον της Ευρώπης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε καλύτερα. Μη μιλάμε για χώρες που ούτε καν γνωρίζουμε. Γίνονται προτάσεις ψηφίσματος και στην ουσία δεν έχουν καμία σημασία, τις πετάμε στο κάλαθο των χρήστων. Κανένας δεν ενδιαφέρεται επί της ουσίας για τα θέματα αυτά. Ε. Σας ευχαριστώ και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Χρήστος, Χρήστος Στυλιανίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμένη αυτή ε, περίπτωση του δικηγόρου και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Λάνι Μασέκο και του συγκατηγορούμενου του Μπέκη Μακούμπου σε αρχισυντάκτη του περιοδικού The Nation. Ήδη από τις αρχές του Μαρτίου 2014 εκφράζαμε τις ε, σοβαρές μας ανησυχίες ε, για την ελευθεροτυπία, για την ελευθερία έκφρασης της Βαζιλάντη. Οι Μασέκο και Μακούμπου συνελήφθησαν στις 17 Μαρτίου του 2014 αφού είχαν γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό The Nation ε, επεκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η δικαιοσύνη έναν θεωρητή σε διαβούλευση με τους εταίρους μας παρακολουθήσαμε από κοινού τις υποθέσεις και ο πρέσβης Μαμπάνε παρακολούθησε τεράστια σύνθεση επαφή με την ομάδα δικηγόρων, με την οικογένεια ε, και επέβαλε επίσημο έτοιμο να επισκεφθεί τους δύο κρατούμενους ε, στις φυλακές. Ε, επίσημη δήλωση της Ένωσης στις 31 Μαρτίου του 2014 ε, υπήρξε επίσης όπου εκφραζόταν η ανησυχία μας για την κράτηση των δύο κατηγορούμενων και τον Ιούνιο του 2014 πάλι στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου ήταν τα, οι εργασιακές συνθήκες της ΟΑΖΑΔΙ επίσης υπήρξε δήλωση όμως παρά τα αυτά καταδικάστηκαν σε διετή κάθριξη οι δύο αυτοί χωρίς να τους ε, δοθεί δυνατότητα να εξαγοράσουν την ε, ποινή τους με χρηματικό πρόστιμο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι άδικα και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει δήλωση εκπροσώπου μετά αυτές τις ε, πολύ σοβαρές ποινές τον Ιούλιο 2014 και τότε ζητούσαμε από τι αρχέ τη ε, Σουαζιλάνδη ε, να σεβαστούν και να προωθήσουν την ε, ελευθερία έκφραση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας, αλλά και οι διεθνεί και περιφερειακέ υποχρεώσει τη χώρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται ότι το ιστορικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι άκρο ανησυχητικό. Δυστυχώ είναι εξαιρετικά βραδία η πρόοδο, όμω ε, Λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν υπάρχει πλέον απαγόρευση για τις συνδικαλιστικέ ενώσει, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι είναι εγγυημένο το ότι οι συναντήσεις τους θα παραμένουν ε, ανενόχλητες, θα γίνονται ανενόχλητα μάλλον. Ε, ούτε εγγυάται κανείς ότι θα απελευθερωθούν οι αγωνιστές συνδικαλιστές. Εμείς επαναλαμβάνουμε και τις πιέσεις που δέχεται ο δικαστικός κλάδος Ο Ραμοπιτέτη, Γενικός Αγγελέας, κατηγορείται για 28 παραβιάσεις και για κατάχρηση εξουσίας μεταξύ άλλων. Ο δικαστής Μελάν ε, που δίκασε τους δύο αυτούς ε, είναι ο ίδιος τώρα, ε, κρατείται ο ίδιος και για αυτός λόγω κατάχρησης εξουσίας. Και τέλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρακαλώ Ησυχία, λέει ο πρόεδρος. Ολοκλήρωσε όμως ο Επίτροπος εν τω μεταξύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος. Από το Ευρωπαϊκό Λεκόμα, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, την Άλντε, την ECR, συντηρητικούς του μεταρρυθμιστές την ε, Γκουε, τους πράσινους και την EFFD. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και ψηφίζουμε αμέσως μετά. colleagues, We will begin the votes in one minute's time. So one minute, please. Αγαπητοί σε ένα λεπτό ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Γι' αυτό παρακαλώ να πάρτε τις θέσεις σας αμέσως.